przewodniczący! E, witam jeszcze raz koleżanki i kolegów. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Πριν όμως από αυτό, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Γιάννος Βοησεχόφσκι, ο οποίος έχει ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Γιάννος Βοησεχόφσκι. Ε, κύριε Πρόεδρε, ε, υψηλή προσκεκλημένη. Ε, χθες στην Πολωνία, στο Woods, ε, σε χώρο εργασίας, σε ένα γραφείο, Ξαναξεκινάω όμως. Κύριε Πρόεδρε, εχθές στην Πολωνία, στο Γουτς, σε ένα γραφείο ενός βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δολοφονήθηκε ένας βοηθός, ο βοηθός μου. Αυτό ήταν κρατικό έγκλημα και ο εγκληματίας είπε ότι μισεί το κόμμα του δικαίου και της δικαιοσύνης και ε, αυτό οδήγησε σε αυτή την τραγωδία. Ε, Γενικώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να καταδικάζει τη βία διότι στην πολιτική και στην Ευρώπη δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για τη βία και θα παρακαλούσα να κρατήσετε ενός λεπτού σιγής ε, για το άτομο αυτό το οποίο δολοφονήθηκε σκληρά μέσα στο γραφείο ενός Ευρωβουλευτής. Παρακαλώ να σηκωθείτε όλοι. Madame, the floor is yours. 664. 684. Yes. για για voorzitter. Voorzitter, dank. Το 684 έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι μόλις δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μόλις δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. είδαμε ότι κάποιοι μας έλεγαν να ψηφίσουμε κάποιες αποφάσεις, μετά κάποιοι άρχισαν να μπαίνουν στο κοινοβούλιο με μπαλόνια. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό ε, περιποιεί τη στο κοινοβούλιο, κύριε Πρόεδρε. Περνάμε κυρίε και κύριοι στην ψηφοφορία. Σας παρακαλώ να περάσουμε αγαπητοί συνάδελφοι στην ψηφοφορία. Bye. Σας παρακαλώ, βλέπετε ότι υπάρχουν μπαλόνια. Θα πρέπει να αποφασίσετε είναι νόμιμο ή όχι να βρίσκονται μπαλόνια μέσα στο ημικύκλιο. Μπορούμε να φέρουμε και εμείς ε, πορτοκαλί και μόβ. Ε, είναι πολύ ωραία. Ε, μπορούμε να σας τα φέρουμε και εμείς αυτά μπαλόνια την επόμενη φορά, αν επιτρέπετε. Dear colleagues, we Πρόεδρος, αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα θα ψηφίσουμε για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Αυτό ακριβώς το ζήτημα σχετίζεται και με τα μπαλόνια αυτά, με αυτή την επίδειξη αν θέλετε. Επειδή λοιπόν η ψηφοφορία αυτή θα λάβει χώρα σε 40 περίπου λεπτά, σας παρακαλώ ως έτσι μια καλή κίνηση, μια χειρονομία καλή ε, για όλους εμάς, σας παρακαλώ να βγάλετε τα μπαλόνια από το ημικύκλιο τη Ολομέλεια. Σας παρακαλώ. Βέβαια η απόφαση είναι δική σα, σα παρακαλώ πάντω. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, μόλι ξεκινήσαμε την ψηφοφορία. Όπως προβλέπει λοιπόν η μερίσια διάταξη θα ψηφίσουμε με βάση την απλουστευμένη διαδικασία την έκθεση του κυρίου Ρανζέλ για την αναθεώρηση τη Συμφωνία Πλησίου για τι σχέσει μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Επιτροπή. Πρόκειται για σημαντικότατη ψηφοφορία. Έχουμε μία και μόνη ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ευχαριστώ πολύ. Εγκρίθηκε η έκθεση. Όπως προβλέπει η μερίσια διάταξη, τώρα ψηφίζουμε τι εκθέσει του κ. Ρουανζέλ για την προσαρμογή του κανονισμού του Κοινοβουλίου στην αναθεωρημένη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Θέτω σε ψηφοφορία την έκθεση. Εδώ πρέπει να υπάρχει ειδική πλειοψηφία, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Υπάρχει ειδική πλειοψηφία, επομένω εγκρίνεται η έκθεση αυτή του κυρίου Ρανζέλ. Θα ήθελα να αναφέρω ότι πρόκειται για τον καρπό μακρών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή κύριο Ρανζέλ αλλά και τον κύριο Λάιν που εξ ονόματός μας ε, ήταν υπεύθυνη για τις διαπραγματεύσεις ε, με την Επιτροπή Σβόποτα, Γουόλις, Hans, Ροτ Μπέρεντ, Ρανζέλ. Όλοι αυτοί οι συνάδελφοι έχουν ε, μια πολύ μεγάλη συμβολή στο αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αυτών. Τους ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, κύριο Μπαρόζο, και τον κύριο Σεύκοβιτ. Νομίζω ότι επιδείξαμε όλοι ανοιχτό πνεύμα. Είναι εξαιρετικό το αποτέλεσμα. Εξού λοιπόν συγχαίρω και τι δύο πλευρέ που καταφέραμε να συνεργαστούμε με επικοδομητικό τρόπο. We are, going to sign the... Και τώρα θα υπογράψουμε την ε, συμφωνία. Κύριε Πρόεδρε, σα καλώ να έλθετε μαζί μου. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε στην ψηφοφορία σειράς εκθέσεων για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Προβλέπει η μερίσια διάταξη την ψηφοφορία της εκθέσεως της κυρίας Γκρέσλε και την έκθεση Ριβελίνη. Την έκθεση Γκρέσλε Ριβελίνη. Πάμε λοιπόν στην αναθεώρηση αυτή του κανονισμού, του σχεδίου κανονισμού. Λοιπόν, ψηφίζουμε την ομάδα 1 πρώτα απ' όλα. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ αυτής της συμβαστικής προτάσεως κατά αποχές εγκρίνεται ψηφίζουμε την πρόταση που τροποποιήθηκε της Επιτροπής ποιος είναι υπέρ κατά αποχή εγκρίνεται ψηφίζουμε το σχέδιο του νομοθετικού κειμένου με ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινά τώρα, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Όπως το διαπιστώνετε κι εσείς, με συντριπτική πλειοψηφία. Συγχαρητήρια λοιπόν στην κυρία Γκρέσλε και στον κύριο Ριβελίνη και σε όλους εκείνους που συνέβαλαν στις διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα. Συγχαρητήρια, εγκάρδια. Τώρα, στην ημερήσια διάταξη, έχουμε την έκθεση του κυρίου Ροπκάη. Τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εξετάζουμε λοιπόν αυτό το σχέδιο κανονισμού. Έχουμε 42 ε, τροπολογίες. Ψηφίζουμε την 1 ως 42. Όλο, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την πρόταση την τροποποιημένη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σχέδιο του νομοθετικού κειμένου με ψηφοφορία που άρχεται τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με συντριπτική πλειοψηφία συγχαρητήρια στον κύριο Ράπκαη, τον εισηγητή μας. Τρίτη έκθεση του κυρίου Γκουαλτιέρη και του κυρίου Σουριάν. Ψηφίζουμε λοιπόν αυτήν την έκθεσή τους όσον αφορά τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 6 κάθετος 2010. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια λοιπόν στον κύριο Γκουαλτιέρη και στον κύριο Σουριάν. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε την οθετική διαδικασία που συνδέεται με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα πολλούς που παρευρίσκονται σε αυτή την αίθουσα. συγχαρητήρια για το έργο τους. Ήταν πολύ πεθυνό το έργο τους, κυρίως οι πρόεδροι των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνέβαλαν στην προσπάθεια. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι πρόεδροι για την έξοχη δουλειά που κάνατε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά και κάποιους που εξεπροσώπησαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις διαπραγματεύσεις Λοιπόν, θα πρέπει να αναφερθούν τα ονόματά τους. Herman Brock, Guy Verhofstadt, Roberto Gualtieri, Ingerbord eh, Gressler, Crescencio Rivellini, Bernard Rapkay. Λάσλο Σουριάν και Συντόνια Γενζογεύσκα που ασχολήθηκαν με τον προπολογισμό αναφέρω αυτά τα ονόματα διότι η δουλειά τους ήταν, το έργο του ήταν τεράστιο για να καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Πιστεύουμε ότι αυτή η συμφωνία θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Συγχαίρουμε όλους αυτούς. Συγχαίρουμε και τη Λέδη Άστον και όσους διαπραγματεύτηκαν εκ μέρους της. Συγχαίρουμε το Συμβούλιο τον κύριο Κριστόφερσεν, τον πρέσβη, που είναι εδώ παρόν, που προετοίμασε τις διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, επιτρέπετε να χειροκροτήσετε τώρα. Where's, where's uh, yes, I prepared some flowers. Έχω ετοιμάσει λίγα λουλούδια για τη Lady Άστον, αλλά δυστυχώς δεν παρίσταται. Ο συνήθως είναι ανάγκη να περιμένουμε τις κυρίες. Ήταν κάτι που δεν είχα προβλέψει, αλλά πρέπει πάντοτε να προσαρμοζόμαστε. Όπως πρέπει να προσαρμοζόμαστε σε όλες τις συνθήκες και να αναμένουμε τα πάντα. Έφτασε.